Το πώ ε, θα εφαρμοστεί τώρα θα το δούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτού του σημείου και πηγαίνουμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή την έκθεση του κυρίου Ριβελίνη για την απαλλαγή 2009. Και δίνω αμέσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Ριβελίνη. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύβο ερήφθη. Με αυτή τη φράση που ε, υπόθηκε όταν ε, διαβήκαμε τον ε, Ρουβίκονα θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Αυτή η παράθεση σηματοδοτεί τότε, ε, και όπως και σήμερα, μια χαρακτηριστική αποφασιστική στιγμή. Ένα πραγματικό ορόσημο στην ιστορία αυτής της θητείας και αυτού του Κοινοβουλίου. Και μέσω της εξουσίας ελέγχου για όλα τα κοινοτικά όργανα και την εξουσία επί του προπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει και επιβάλλει τις αρμοδιότητες της, ε, συγγνώμη, της πολιτικές του προτεραιότητες. Το να τα στερηθεί αυτά θα σήμαινε να κενώσουμε το νοήμα τους το, την αρχή της δημοκρατίας και την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Αυτό που το οποίο συζητάμε τώρα δεν είναι η διεκδίκηση ενός προνομίου, δεν είναι όπως θα ήθελε το Συμβούλιο η διεκδήλωση της βούλησης να αποσπάσουμε με τη βία και να ιδιοποιηθούμε πολιτική εξουσία εις βάρος κάποιου άλλου. Περισσότερο αποτελεί την επιβεβαίωση της, ε, του νόμου νόμιμου και παραβίαση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο καθήκον του να εξασφαλίζει την μόνιμη παρακολούθηση των δαπανών στις οποίες προβαίνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και του δικαιώματός του να αναγνωρίζεται ως αρχή της, της απαλλαγής. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι ένα κύρος το οποίο είναι αυτό αυτό είναι ε, αντιπροσωπευτικό του ε, ευρωπαϊκών λαών Πρόκειται για τη διάρθρωση σε μια οδό. Από τη μια πλευρά υπάρχει μια πρώτη φάση λογιστικής φύσης που αντιπροσωπεύεται από το κλείσιμο των λογαριασμών που βρίσκει που κορυφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 319 της συνθήκης στην χορήγηση απαλλαγή στην Κομισιόν. Και από την άλλη αναπτύσσεται η πολιτική ε, αξία της απαλλαγή, δηλαδή η κρίση που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαχείριση των λογαριασμών του συνόλου των θεσμικών οργάνων άνευ Με μεγάλη δυσαρέσκεια αναγνωρίζουμε ωστόσο πως πολλές φορές έχουμε μπει στην άκρη, πολλές φορές έχει ε, παρεμποδιστεί λειτουργία μας λόγω της ε, ισχνής συνεργασίας ε, που, από πλευράς του Συμβουλίου που συχνά δεν θέλει να συμμετέχει στην ανταλλαγή γράφων και δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητά μας για την απαλλαγή. Γι' αυτούς τους λόγους ε, είμαστε αρνητικοί εντόνως όσον αφορά την εκτέλεση των δαπανών του Συμβουλίου και, να, και είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε την άρνηση της απαλλαγής. Για αυτή τη τελευταία φάση θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε σήμερα, σεβόμενοι τις διαφορετικές απόψεις αλλά και με μοναδικό στόχο να επιβεβαιώσουμε την ολοκλήρωση της Ευρώπης που με μια λέξη γίνεται τελικά η Ευρώπη των λαών. Γι' αυτό και πιστεύουμε και το πιστεύουμε σταθερά ότι η ίδια η Ευρώπη ακριβώς λόγω του χιλιετιών πολιτισμού, λόγω, λόγω του ότι, είναι, ότι πρόκειται για κοινή μοίρα ε, να αντιπροσωπεύουμε την ελπίδα ενός πόλου αναφοράς για έναν κόσμο χωρίς ψυχή που είναι κενό από λόγω του μερκαντιλισμού και σχηματίζεται από τους λαούς μέσα σε μια παράλογη υποχώρηση. Η συνθήκη όμως της Λισαβόνας μας έχει εξασφαλίσει έναν υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας και μας έχει αποδώσει μεγάλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στο σεβασμό της δημοκρατίας και της διαφάνειας που αποτελούν τα θεμέλια του συστήματος προστασίας της Ευρώπης ε, απέναντι στους πολίτες της. Και ακριβώς σήμερα με σεβασμό αυτών των αρχών θέλουμε να μιλήσουμε για τη λειτουργία του Συμβουλίου. Δεν έχουμε κανένα κανένα λόγο λόγο να φοβόμαστε μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ούτε φοβόμαστε την, ε, το διακυβερνητικό θεσμό. Σας ζητώ να ολοκληρώσετε, έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας κύριε Ριβελίνη. Μάλιστα, να κλείσω ζητώντας λοιπόν από ολόκληρο το Κοινοβούλιο να ψηφίσει κατά της απαλλαγής του Συμβουλίου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Το λόγο έχει τώρα Επίτροπος Νταλή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή ε, σημειώνει τη σύσταση του Συμβουλίου να μην χορηγηθεί απαλλαγή στο Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2009. Ε, η Κομισιόν εκφράσει τη λύπη τη ε, για το γεγονό ότι τα δύο σκέλη τη αρχή επί του προπολογισμού δεν κατάφεραν να βρουν μια λύση στην διαφορά αυτή, η οποία συνεχίζεται εδώ και τριετία. Η Κομισιόν ελπίζει ότι το ζήτημα της απαλλαγής του Συμβουλίου θα ρυθμιστεί τάχιστα κατά τρόπο που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ε, διοργανικής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, καταρχάς εκ μέρους του ΕΛΚ, κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, χαιρόμαστε γιατί θεωρούμε σημαντικό να ανταλλάσσουμε απόψεις. Εδώ πέρα μπροστά μας έχουμε το Corpus Delict. Έχουμε τις 34 ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού προς το Συμβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009. Και σας υπενθυμίζω πως θέσαμε άνω των 200 ε, ερωτήσεων και απαντήσατε κάτι παραπάνω από το 10%. Επίσης, Ξέρετε πως το θέμα το οποίο με απασχολεί εμένα είναι το πώς ε, μπλέκονται οι δαπάνες, οι καθαρά διοικητικές εξωτερικής υπηρεσίας με τις δαπάνες της εξωτερικής πολιτικής. Κοιτάξτε, τα επόμενα χρόνια θα προχωρήσουμε πιο κοντά σε μια λύση αν βρεθεί λίγη καλή θέληση και απευθύνω έκκληση κύριε Πρόεδρε γιατί θεωρούμε πως ε, από την Ουγγρική Προεδρία και μετά έχουμε μόνο βήματα προς τα πίσω. Η μεγαλύτερη πρόοδο σημειώθηκε επί Ισπανικής Προεδρίας Πρέπει λοιπόν ε, να σας υπενθυμίσουμε πως το Κοινοβούλιο είναι αρχή της απαλλαγής του προπολογισμού. Δεν είναι δυνατόν να παραιτηθούμε από τα δικαιώματα που έχουμε, τα οποία δεν είναι και τόσο πολλά. Θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν να ε, απαιτήσουμε να σεβαστούμε τα, να σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Ε, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αμοιβαιότητα, δεν είναι δυνατόν υπάλληλοι του Συμβουλίου να μην δίνουν λογαριασμό στο Κοινοβούλιο. Θε, απαιτούμε περισσότερη καλή θέληση από αυτή η οποία έχει επιδειχθεί μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ κύριο Γκαΐρ για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της απαλλαγής του Συμβουλίου αποτελεί θέμα αντιπαράθεσης εδώ και χρόνια μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η διαδικασία όπως το ερμηνεύουμε εμείς, ε, προκύπτει από το άρθρο 319 περί απαλλαγής του Συμβουλίου και τις ανάλογες παραγράφους του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη το Συμβούλιο και θεωρεί πως μπορεί, εφόσον χρησιμοποιεί τμήμα του προπολογισμού της Κομισιόν, να λαμβάνει απαλλαγή μαζί με την ε, Κομισιόν. Εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού τα έχουμε πει πολλές φορές. Απλά θα πω πως ε, αυτά τα οποία ακούστηκαν πολλά και δεν ήταν συνεκτικά. Τώρα φαίνεται πως το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο γενικών γραμματέων, το οποίο ε, θεωρώ πως δεν έχει αρκετά ε, μεγάλη πολιτική εντολή να διαπραγματευτεί μαζί μας για την ε, απαλλαγή του Συμβουλίου. Και θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για αυτή του την προσφορά. Θεωρώ πως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την προσφορά διαπραγματεύση με μια υψηλού επίπεδου διαπραγματευτική ομάδα και να μην ε, επιβαρύνουμε εκ των προτέρων αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό το οποίο προτείνω στην ομάδα μου είναι αποχή. Τον λόγο... Θέλετε, Θέλετε κύριε Γκέρ προφορική ερώτηση με το ύψωμα της μπλε κάρτας. Ευχαριστώ. κύρια Πρόεδρε, ναι, συμφωνούμε εδώ πέρα στην ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θέλουμε να συστήσουμε να μην δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Οπότε θέλω να ακούσω εάν εξακολουθεί να έχει αυτή την άποψη η Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα γιατί δεν ήταν σαφές. Υπάρχουν φήμες εδώ πέρα πως σοσιαλδημοκράτες αποφάσισαν να αλλάξουν θέση και να υπερψηφίσουν την απαλλαγή. Θέλω να μου πείτε εάν ισχύει κάτι τέτοιο και εάν ναι, γιατί η σοσιαλδημοκρατική κοινοβουλευτική ομάδα μετέβαλε άποψη. Υπάρχουν φήμες που λένε πως αυτό σχετίζεται με τον νέο πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θέλω να μου απαντήσετε όμως εσείς. Ευχαριστώ να απαντήσω. Είναι φήμες. Και θα μπορούσα να πω πως δεν σχολιάζω φήμες, αλλά ούτως ή άλλως μόλις παρουσίασα τη θέση της ομάδας μας, η οποία είναι αποχή σε αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα είναι προδικασμένο εκ των προτέρων. Το είπα. Τα υπόλοιπα ήταν φήμες. Σας ευχαριστώ. Είναι σαφές. Τον λόγο έχει ο κύριος Χιλακάκης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του Γενικού Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, η διοίκηση του Συμβουλίου οφείλει να υπόκειται σε δημοκρατική λογοδοσία προς τους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης και να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση του Συμβουλίου επί πολύ καιρό δεν αποδέχθηκε καμία πρόσκληση για να συναντηθεί με την κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρμόδια για την διαδικασία της απαλλαγής και η οποία ακόμη δεν έχει λάβει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει θέσει. Οι Ευρωπαίοι πολίτες όμως δικαιούνται καλύτερη ενημέρωση σχετικώς με το πώς δαπανούνται οι φόροι τους. Θεωρώ λοιπόν πως δεν πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή και αν αποτύχει και η τελευταία προσπάθεια διαπραγμάτευσης και στη περίπτωση που το Συμβούλιο συνεχίσει να έχει διαφορετική νομική άποψη σε σχέση με τις δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου για το θέμα και με δεδομένο ότι ο διάλογος έχει ως τώρα καταλήξει σε αδιέξοδο και η νομική εκκρεμότητα εκθέτει όλους τους εμπλεκομένους θεσμούς, έχουμε πλέον μία μόνο δυνατότητα, την παραπομπή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε να ξεκαθαρίσει άπαξ και διαπαντός αυτό το θέμα και να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική θεσμική λειτουργία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σκυλακάκη. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαρνέσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ο φίλος κύριος Ριβελίνη τα είπε όλα δεν είναι ο Κέσαρας τώρα στο Κοινοβούλιο, ήταν ο Ρουβίκονας και η δέλευσή του ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, αλλά τον έχουμε διαβεί και έχουμε διαβεί και το Ρήνο στο μεσοδιάστημα. Ουσιαστικά παίζουμε το ίδιο παιχνίδι, το παιχνίδι της εξουσίας. Ε, ποιος έχει τη μεγαλύτερη εξουσία, το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Όσοι ήμασταν βουλευτέ και στην προηγούμενη θητεία βλέπουμε ότι το ίδιο παραμύθι επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δίχως τέλος είναι αυτό. Το Συμβούλιο δεν έχει αναγνωρίσει πλήρως ε, τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα εδώ σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλεγχο, είναι πολύ σημαντικέ οι εξουσίε αυτέ. Ε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε λοιπόν τη χωρί απαλλαγή. Ευχαριστώ. Κύριο Στάς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Όπως και η κυρία Γκρέσλε, χαίρομαι για το ότι είναι παρόν το Συμβούλιο. Ε, είδα όμως τον πίνακα των ομιλητών και βλέπω πως δεν ζητήσατε το λόγο. Νομίζω πως θα πρέπει στο τέλος της συζήτησης να αντιδράσετε στις παρατηρήσεις μας. Ε, κύριε Στάς βεβαίως θα λάβουν το λόγο και θα απαντήσουν ε, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Α, εντάξει, γιατί δεν ήταν στον κατάλογο λέει ο κύριος Στάς. Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία τραβάει εδώ και τρία χρόνια και είναι άσχημη αυτή η υπόθεση. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Δεν συμβαίνει αυτό. Είναι άκαμπτο το Συμβούλιο και ακούγονται πράγματα για μια συμφωνία κυρίων ε, που έκλεισε πριν από 40 χρόνια. Είχε συναυθεί. Εντάξει, συμφωνία κυρίων, αλλά δεν συμφέρει φέρεστε ως κύριοι, κύριοι του Συμβουλίου. Τι ζητάμε εμείς λοιπόν. Να δώσουμε απαλλαγή στον προπολογισμό του Συμβουλίου όπως γίνεται και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Τόσο φοβερό είναι. Τα λεφτά τα οποία δίνει ο φορολογούμενος να μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αυτό είναι το ζήτημά μας. Η ομάδα μας, η πράσινη και η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δεν θα δώσουν απαλλαγή στο Συμβούλιο. Γιατί θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως πρέπει να ξοδεύονται σωστά τα χρήματα. Κανείς δεν λέει στη συζήτηση πως κάνει απάτη το Συμβούλιο. Κανείς δεν λέει πως έχει υπάρξει κάποια παρατυπία. Είναι ζήτημα απλά δημοκρατικού ελέγχου από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που είναι το καθήκον της. Η μόνη απάντηση που λάβαμε ήταν μια επιστολή της Δευτέρας Ιουνίου όπου λένε κοιτάξτε να δείτε εμείς ερμηνεύουμε αλλιώς τη συνθήκη οπότε θεωρούμε πως αν δίνεται απαλλαγή στην Κομισιόν ε, έχει τελειώσει το όλο ζήτημα. Ε, όχι, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, δεν μπορείτε σοβαρά να ισχυρίζετε κάτι τέτοιο. Πρώτον, πρόκειται για τακτική ετών και δεύτερον, δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε αυτή την ερμηνεία, μπορούμε να τα ακολουθήσουμε για οποιοδήποτε θεσμικό όργανο. Δεν είναι δυνατόν. Ή αλλιώ θα έπρεπε να εμφανίζεται το Συμβούλιο ενώπιον τη ε, Κομισιόν. Και σβήνει το μικρόφωνο του κυρίου Στά. Δίνω τον λόγο στον κύριο, κ. Σόντεργαρντ. Δεν έχει. Σας ευχαριστώ. Ε, υπάρχει εδώ πέρα μια ξεκάθαρη και ομόφωνη θέση μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή στο Συμβούλιο. Τα πράγματα δεν είναι καινούργια αυτά. Ήδη από το 2009 αναβάλουμε την απαλλαγή, την αναβάλαμε τότε για το φθινόπωρο και μετά δόθηκε μια απαλλαγή γιατί έκανε κάποιες παραχωρήσεις το Συμβούλιο. Όχι πολλές, αλλά εν πάση περιπτώσει προς τη σωστή κατεύθυνση. 2010 το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς συνέβη. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα όπως ακούσαμε. Αρνείται, εξακολουθεί να αρνείται να απαντήσει τις ερωτήσεις μας το Συμβούλιο. Πώς μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή όταν δεν λαμβάνουμε απάντηση στις ερωτήσεις μας. Δεν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να το κάνουμε αν έχουμε αυτοσεβασμό. Οπότε πραγματικά λυπούμε ειλικρινά για το ότι η πλειοψηφία των σοσιαλιστών και δημοκρατών άλλαξε στάση και λυπούμε για το ότι δεν έχουμε ενότητα στην Επιτροπή Ελέγχου του Υπερυπολογισμού. Θέλει να μείνει μόνο του, μόνο της η σοσιαλδημοκρατική ομάδα. Υπάρχει όμως νομίζω εδώ μέσα μια πλειοψηφία υπέρ της διαφάνειας. Η κυρία είναι για 1,5 λεπτό. Η έγκριση της διαχείρισης ε, των χρημάτων των φορολογουμένων, η διαδικασία της απαλλαγής δηλαδή που χορηγεί το Κοινοβούλιο στα θεσμικά όργανα έχει γίνει αστείο τελικά. Το μεγαλύτερο μέρος ε, του προϋπολογισμού κάθε χρονιά πλέον ε, αυτό το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κομισιόν είναι γεμάτο από παρατυπίες παρόλα αυτά με τα χαράς χορηγεί το Κοινοβούλιο απαλλαγή και την ε, αστυνομική ακαδημία θα χορηγήσουμε απαλλαγή φέτος παρότι υπήρξαν ε, καταχρήσεις ε, πολύ σημαντικές το 2009. Όταν όμως μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αρνείται το Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή, παρότι δεν υπάρχει καμία επίκριση σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση του θεσμού αυτού. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η ασυνέπεια. Πολύ απλά πρόκειται για παιχνίδια εξουσίας. Το ε, Κοινοβούλιο νομίζω ότι έτσι θα δείξει τη δύναμή του. Ε, αλλά τελικά ε, δείχνει ε, ότι παραγνωρίζει τα χρήματα των φορολουμένων που υποτίθεται ότι ε, σέβεται και βλέπουμε ότι τελικά ε, μόνο αυτό εγκρίνει μόνο του λογαριασμού του και αυτό υπάρχει, στο σημείο αυτό υπάρχει σύγκρουση ε, συμφερόντων. Είδαμε κάποιες εκθέσεις προηγούμενη εβδομάδα από τους ε, ελεγκτές που δεν ε, δείχνουν ότι είναι άσπλα τα πράγματα. Εγώ έχω ψηφίσει κατά της απαλλαγής ε, ε, της επιτροπή του Κοινοβουλίου, θα ψηφίσω και κατά της απαλλαγής του Συμβουλίου, από τη στιγμή που δεν μπορώ να είμαι βέβαιο ότι έχουν δαπανηθεί σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ πολύ. Χολμάγερ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πρώτα απ' όλα, σε αντίθεση με την προηγούμενη ομιλήτρια, να ξεκαθαρίσω πως όσον αφορά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ δεν θέλω να πω πως υπάρχει κάποια δυσπιστία εδώ πέρα προς το Συμβούλιο ή ότι υποθέτουμε πως έχει υπάρξει κάποια παρατυπία στα έξοδα. Αλλά εμεί θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και των τριών θεσμικών οργάνων. Να σας πω, κοιτάξτε, ε, είμαι και η εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Υπάρχουν ε, σαφή πλεονεκτήματα λοιπόν στο να συνεννοηθούμε για αυτό το θέμα, γιατί έτσι θα μας ευχαριστούν οι φορολογούμενοι. Το να συντονιστούμε δηλαδή και να μην ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον ε, άλλον. Και, και όσον αφορά τα κίνητα και όσον αφορά τους διερμηνείς και τα Τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να μην α, υπάρχει αυτή η στάση, αλλά να απαντάμε τουλάχιστον τις ερωτήσει ο του άλλου. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Τι μας ζητούν ε, οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, καλύτερο είναι ο εχθρό του καλού τελικά σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι έχουμε ακολουθήσει λάθο δρόμο και βλέπω ότι και οι δύο τροπολογίε του κυρίου Ριβελίνη ε, εύγλωτε είναι διότι ουσιαστικά μα πηγαίνουν πίσω στι ε, πρώτε προτάσει ε, και πραγματικά είναι πάρα πολύ ψοκίνδυνο αυτό κατά την άποψή μου. Οι Σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες συζητήσαμε σε βάθο το θέμα, απαιτούμε διαφάνεια, απαιτούμε να είναι όλα ξεκάθαρα και σαφή. Πάντα το πράταμε, αλλά δεν συμφωνούμε με αυτό το δρόμο που έχει επιλεγεί ε, μια ομάδα υψηλού επίπεδων δύο θεσμικών οργάνων, όπω πρότεινε ο συνάδελφο Γκάγκερ, νομίζω ότι είναι ο σωστότερο δρόμο που δείχνει οριμότητα. Εσά, κυρία Γκρέστερ, δεν σα αρέσουν οι υπάλληλοι. Εγώ νομίζω ότι κάνουν σωστά την ε, δουλειά τους και το να δώσουμε στην, ε, στο δικαστήριο τον τελευταίο λόγο είναι λυπηρό. Νομίζω ότι απαιτείται μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Άσβορθ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Σύμφωνα με την Διοργανική Συμφωνία του 2005, το Συμβούλιο προέδισε συμφωνία με αυτό το Κοινοβούλιο και δεν είναι αποδεκτό πολλά κράτη-μέλη να εξακολουθούν να αγνοούν αυτές τις δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα, υπό το φως της συνθήκης Λισαβόνας, πρέπει πλέον να συνειδητοποιήσουν την υποχρέωση για να η καλύτερη συνεργασία με, αυτή, με αυτό το σώμα. Το Συμβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του. Δεύτερον, Παρακαλώ τόσο το Συμβούλιο όσο και την Κομισιόν να κατανοήσουν ότι οι διαρκείς παρατηρήσεις και ο έλεγχο και αντιπαράθεση με το Συμβούλιο, με το ελεγκτικό συνέδριο είναι ιδιαίτερα βλαβερό και ζημιώνει την εικόνα μας προς το ευρύ κοινό. Δεν αρκούν οι τεχνικές εξηγήσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σαφείς δράσεις να πούμε το, ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν πρέπει να δώσουν πιο επίγοντα χαρακτήρα στην επίτευξη ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας. Merci. Κυρία Μακοβέη, σας ευχαριστώ. Το Συμβούλιο δήλωσε πως η διαδικασία απαλλαγής 2009 θα έπρεπε, έχει ήδη ολοκληρωθεί όταν δόθηκε απαλλαγή στην Κομισιόν. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορώ να πιστέψω πως το Συμβούλιο θέλει να δαπανίσει χρήματα χωρίς δημοκρατικό έλεγχο. Ωστόσο αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Δεν είναι ότι υπεύθυνο αυτό, ούτε παράδειγμα χρηστή διακυβέρνησης, διαφάνειας ή λογοδοσίας. Είναι αυτό ιδιαίτερα πιο ανησυχητικό κατά τη διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης και της κρίσης εμπιστοσύνη όπου πρέπει να δώσουμε λογαριασμό για κάθε ευρώ και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Έχουμε το δικαίωμα να ελέγχουμε το εκτελεστικό και τις δαπάνες του. Το, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απομακρυνθεί από αυτή την πρακτική και γι' αυτό και στηρίζω απόλυτα τη θέση του εισηγητή για την μη χορήγηση απαλλαγής στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μακοβέη, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Λιμπεράτσκι για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Γκάιερ παρουσίασε την θέση των σοσιαλδημοκρατών για αυτό το θέμα, καθώς και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ακολουθεί την αρχή του σεβασμού της ισορροπίας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τονίζουμε ακόμα μια φορά τη σημασία της διαφάνειας για τα οικονομικά θέματα, τα δημοσιονομικά θέματα και είμαστε της άποψης να ζητήσουμε από το Κοινοβούλιο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες μας στην ε, δημοκρατικό έλεγχο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ιστορική στιγμή όπου κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος θα πρέπει να ελέγχεται ε, και γι' αυτό και ανησυχούμε για την τάση αυτή του Συμβουλίου, την απροθυμία δηλαδή να προβεί σε ανοιχτό διάλογο ανεξάρτητα από το πολιτικό του χρωματισμό. Κατά τη λοιπόν υπάρχει μάλλον κάποιο διοικητικό ή γραφειοκρατικό κομμάτι του Συμβουλίου που δεν είναι πρόθυμο να το κάνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Για ένα λεπτό, η κυρία Μπένοβα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, ε, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, συνάδελφοι, νομίζω πως το θέμα που συζητάμε εδώ, εκτός από τις νομικές και θεσμικές του ε, διαστάσεις, έχει και πολιτικές διαστάσεις. Το Κοινοβούλιο έχει κάθε αρμοδιότητα και δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά του, τις αρμοδιότητές του. Και αυτό το κάναμε γιατί το Συμβουλίο δεν συμμορφώνεται προς υποχρεώσεις του. Έχουμε τώρα νομική σύγκρουση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα τη Ένωση, δεν είναι καθόλου καλό αυτό όσον αφορά την νομιμότητα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν εξυπηρετεί την αρχή ε, της αρχές μας αν... Ε, αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους τα θεσμικά όργανα. Έχουμε ένα σωρό άλλα προβλήματα που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τους δικούς μας, ε, τις δικές μας ε, θέλουν να αντιμετωπιστούν τα δικά τους προβλήματα, όχι τα δικά μας. Θα πρέπει λοιπόν να σύντομα να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούλτερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις συνθήκες. Είναι η αρχή χωρίς απαλλαγής των θεσμικών οργάνων, τα οποία λογοδοτούν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για το Συμβουλίο Υπουργών. Μια έσχατη λύση, κατά την άποψή μου, θα ήταν να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι η ιδεώδης λύση. Να τονίσω ότι το Κοινοβουλίο είναι ανοιχτό προς διάλογο με το Συμβούλιο και θα ήθελα ανοιχτά να απευθυνθώ ε, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό και στο πολιτικό επίπεδο ε, να τους παρακαλέσω να έρθουν σε επαφή με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να μην ε, αρνούνται, να εμφανίζονται όπως κάνουν μέχρι τώρα αν το Συμβούλιο εξακολουθεί να αρνείται να ε, έρθει σε διάλογο με την Επιτροπή Ανοιχτού Προβλήσμου, δεν πρόκειται να λύσουμε τίποτα. Ο κύριο Ντάλιτο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε τα διάφορα σχόλια από όλου του βουλευτέ και ακούσαμε κάποιες εκκλήσεις για συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, τις οποίες καλωσορίζουμε η Κομισιόν πρέπει να τονίσει την πολιτική φύση του ζητήματος. Η Κομισιόν θεωρεί πως όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργαστούν για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Θα πρέπει ούτως ή άλλω η αλλω η κομισιον να συνεχίσει την ενεργή συμμετοχή τη στη διαδικασία και μπορώ να δεσμευτώ πώ έχετε οπωσδήποτε έναν καλό συνομιλητή στο πρόσωπο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Υπουργό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η θέση του Συμβουλίου παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την επιστολή της 2ης ε, Ιουνίου και 17ης Οκτωβρίου και το Συμβούλιο θεωρεί πως η διαδικασία της απαλλαγής ολοκληρώθηκε στις 10 Μαΐου όταν δόθηκε απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε τη συζήτηση που υπάρχει και γι' αυτό το Συμβούλιο υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητηθεί μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Συμβούλιο για να υπάρξει μια συμφωνία για την χορήγηση απαλλαγή ε, και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο δημοσιονομικών αρχών και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει γρήγορα να προχωρήσει σε έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία. Δεν έχουμε κανέναν όρο όσον αφορά τη μορφή της εν λόγω συμφωνίας. Όμως θα θέλαμε να τελειώσει η περίοδος της παρεξήσεις και να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο εισηγητής ο κύριος Ρελίν για τη Presidente. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ διαρωτώ με. Αφόσον είναι δικαίωμά μας να δίνουμε ή όχι την απαλλαγή στο Συμβούλιο. Το ίδιο το Συμβούλιο θεωρεί ότι χωρίς καμία συνεργασία είναι ήδη κεκτημένο του Μα τότε τι δικαίωμα είναι αυτό, τι κύρος έχει αυτό το κοινοβούλιο και τι νόημα. Εμείς ε, δεν θεωρούμε πως η θέση μας ε, θα ακυρώσει την συμφωνία των κυρίων και είναι και απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το από Κοινοβούλιο ε, έχει αποφασίσει σε μεγάλη, μεγάλο μερίδιο, δηλαδή ψηφία είναι υπέρ της θέσης μου και καλό και όσους ακόμα έχουν αμφιβολίες να υποστηρίξουν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου που πρέπει να γίνονται σεβαστά. Φυσικά και το εύχομαι ε, μια έκκληση θα κάνω και προς το Συμβούλιο γιατί αν από σήμερα αλλάξει η θέση αν υπάρξει μια πραγματική συνεργασία αν αναγνωρίσει το ρόλο του Κοινοβουλίου ως δημοκρατικού εκπροσώπου των δικαιωμάτων των πολιτών τότε θα επανεξετάσουμε τη θέση μας. Ε, διδικό, έκκληση ε, προς εσάς λοιπόν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η απαλλαγή προς την Κομισιόν στις 10 Μαΐου δεν έχει καμία σχέση. Πρόκειται για δύο, διαφορετικά, ε, δύο διαφορετικούς δρόμους και εδώ πρόκειται για ένα πολιτικό αποτέλεσμα μεγάλης πολιτικής σημασίας στη σημερινή ψηφοφορία. Ε, μια έκκληση λοιπόν, αλλά δεν υπάρξει θετική απάντηση από πλευρά του Συμβουλίου, ζητώ από όλου του συναδέλφου να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αρνούμενοι την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Λιβελίνη. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Θα γίνει η ψηφοφορία σήμερα στις 12.30. Τώρα προβλέπεται η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή και με τα χαράς καλωσορίζω σήμερα τους Επιτρόπους Μπαρνιέ, Νταλή και Κρόους. Το θέμα, το εισόδων των ερωτήσεων είναι ε,